Buongiorno a Καλή σα ημέρα. Και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ε, συνάντησή μας μετά από τις ερηνές διακοπές. Θα ήθελα να αρχίσω ευθύ αμέσω, αφού πρώτα καλωσορίσω και ευχαριστήσω την Επίτροπο Fisher Bowl και το τους ε, συνόδους τους. Ε, θα ήθελα να εγκρίνουμε τη μέσα διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, να μπορούμε να την εγκρίνουμε. Καλημερίζω και τους διερμηνείς ε, Έλληνο Σήμερα έχουμε όλες τις γλώσσες εργασίας. Περνάμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσεως της 21ης ε, Ιουλίου και 29ης Ιουλίου 2009. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι το πέρας της συνεδριάσεώς μας, ε, τα πρακτικά θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Να σας πω επίσης πως η σημερινή συνεδρίαση θα μεταδοθεί μέσω του διαδικτύου Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για τις εργασίες μας μπορεί να την παρακολουθήσει. Και τώρα ξεκινάμε με το πρόγραμμα της κοινή γεωργικής πολιτικής στη διάρκεια της 7 κοινοβουλευτικής περίοδου. Έχουμε τη χαρά να παρευρίσκεται η αρμόδια Επίτροπος Γεωργίας και Ανάπτυξης Πέτρου, κυρία Μαρία Φίσορ που θα παρουσιάσει το πρόγραμμα το οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Θα, με την ευκαιρία αυτή θα μπορέσουμε να εξετάσουμε και κάποια πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν στην κρίση του γαλακτοκομικού τομέα. Είναι κάτι που συζητήσαμε στην τελευταία συνεδρίασή μας και θεωρώ πως θα ήταν ιδιαίτερα σκόπιμο σήμερα να μεταφέρουμε στην Επίτροπο το συνέστημα της Επιτροπής μας και τις εκφράσουμε την, ανησυχία μας σχετικά με αυτήν την δραματική κρίση που αντιμετωπίζει ο τομέας της ο γαλακτοκομικός. Αγαπητή Μαριάν, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχεί για την παρουσία σου σήμερα εδώ και ελπίζω αυτή η παρουσία να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου, κατά τη διάρκεια της οποίας ε, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε σημαντικές αλλαγές της κοινή αγροτική πολιτικής. Η εφαρμογή της ηθίκη Λισαβόνας, εάν το δημοψήφισμα του Οκτωβρίου στην, Λισαβό... στην ε, Ιρλανδία έχει αίσιο πέρα και την ε, περαιτέρω μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής αλλά και τις συζητήσει για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν ε, τους ε, εχθρούς της κοινής αγροτικής πολιτικής, εχθροί οι οποίοι θέλουν να περιορίσουν τον προϋπολογισμό που δίνεται στην κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια ευθύνη, σήμερα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με την μελλοντική κοινοβουλευτική περίοδο που θα είναι η κοινοβουλευτική περίοδος η οποία θα αποφασίσει κατά πόσο θα υπάρξει ή όχι μια αγροτική πολιτική μετά το 2013. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη που φέρουμε και θα πρέπει να παίξουμε ένα ομαδικό παιχνίδι για να καταδείξουμε την σημασία αυτής της πολιτικής όχι μόνο για τους γεωργούς αλλά για όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Επίτροπε, αγαπητή Μαριάν, έχει το λόγο. President, Vice Presidents and Honourable Member of the Agricultural Committee, it's, it's great to... Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ ε, ξανά μαζί σας ε, μετά από ένα καλοκαίρι όπου περάσαμε καλά, ε, ελπίζω. Χαίρομαι που ο Πάολο Ντικάστρο, φίλος μου, είναι, προεδρεύει αυτής της Επιτροπής. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Γι' αυτό χαίρομαι που θα, μπορέσω να, θα μπορέσουμε να μπούμε στο ψητό, αν θέλετε, και να συζητήσουμε ε, τα θέματα μας ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την, ε, για την εκλογή σας και για το διορισμό σας στην Επιτροπή Γεωργίας. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία μου είναι οικία και επίσης βλέπω και άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζω τόσο καλά, δεν είναι, πια, δεν είναι τόσο γνωστά και όμως θα ήθελα να τους γνωρίσω περισσότερο. Επίσης ήθελα να να σας πω ότι θα ήθελα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει στο μέλλον έναν ε, μεγαλύτερο ρόλο στον καθορισμό της ε, ε, ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής. Αρκεί βέβαια και όλα τα κράτη να επικυρώσουν την συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθω αργότερα. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και Ελπίζω να με συγχωρήσετε και ζητώ συγγνώμη σήμερα το πρωί για το γεγονό ότι θα αναφερθώ μόνο σε ορισμένα από τα πολλά αυτά θέματα. Πιστεύω ότι με την παλιά γκρι είχαμε μια τόσο καλή σχέση, εν μέρει επειδή ήμασταν πάντοτε ειλικρινεί μεταξύ μας, σαφής και άμεση στις συζητήσεις μας. Και θα ήθελα να αρχίσω της, ε, τη συνεργασία μας στο ίδιο στυλ, με τον ίδιο τρόπο όπως με την παλιά κομμαγκρή, με, την, ε, με το παλιό καθεστώς. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσουμε απόλυτη σαφήνεια τις απόψεις μας, ε, τις απόψεις της νέας Επιτροπής, της νέας Κομισιόν, ιδίως των νέων μελών. Ορισμένοι από εσά τα ξέρετε ήδη τις βασικές ιδέες. Ε, Έχοντα υπόψη τα γεγονότα αυτού του καλοκαιριού, θα αρχίσω καταρχάς με τα προβλήματα του γαλακτοκομικού τομέα έχω επανειλημμένως πει ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και είναι σαφές ότι πρέπει να δείξουμε να είμαστε μεγαλόψυχοι και να δείξουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τις ενέργειες που θα κάνουμε αλλά πιστεύω ότι όλοι συμφωνείτε ότι ναι μεν μεγαλόψυχοι, και να δείξουμε κατανόηση βεβαίως αλλά όχι μόνο για να λύσουμε τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα, αλλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή μας για την πολιτική μας με ε, μεγάλη σοφία, μεγάλη προσοχή, μη παραγνωρίζοντας ε, τις προπτικές του μέλλοντος. Να κοιτάμε ε, κοντά μεν, αλλά όχι χωρίς να αγνοούμε το μέλλον. Πρέπει λοιπόν ε, και πάλι να συζητήσουμε το θέμα των ποσοστώσεων γάλακτος ως εργαλείο εγγύησης του μέλλοντος του τομέα. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την αντίληψη. ή Το μέλλον των ποσοστώσεων είναι σαφές ότι θα καταργηθούν το 2015. Αν δείτε όμως την κατάσταση του 2008, έχουμε λιγότερο από το 1 πέμπτο των γαλακτοπαραγωγών που έχουν μείνει μέσα στο σύστημα, ακόμα και αν το σύστημα αυτό είναι διαθέσιμο. Είναι λοιπόν σαφές ότι όπως έχει συμφωνηθεί το 2015 θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις και το σύστημα ποσοστώσεων γάλακτος. Είναι αυτό, αυτή μια απόφαση την οποία ε, χαράξαμε, ένας χάρτης που χαράξαμε το 2003 στην ε, μεταρρύθμιση και το έχω, την, έχει περάσει από, το τσεκ, ε, από τον έλεγχο υγείας της ΚΑΠ και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών χωρών έχουν επιβεβαιώσει αυτή την απόφαση διότι έχουν βάσιμους λόγους που θα τηρήσουν αυτή την απόφαση. Τώρα, μία, ε, ένας κεντρικός προγραμματισμός του συστήματος ποσοστώσεως δεν θα είναι επιτυχής, δεν θα δομήσει σωστά για το μέλλον το γαλακτοκομικό τομέα. Θα μειώσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, θα αυξήσει το κόστος παραγωγής και θα δυσκολέψει τη ζωή στους νέους αγρότες για να επιβιώσουν σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι η σωστή συνταγή αυτή η ε, βαριά, η ε, κεντρική διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να δράσουν οι ενδιαφερόμενοι. Γι' αυτό έχω, τους έχουμε πει στους γαλακτοπαραγωγούς να προετοιμαστούν για ένα μέλλον χωρίς ποσοστώσεις. Και αν τώρα οπισθοχωρήσουμε και οπισθοδρομήσουμε θα δημιουργηθεί χάος και τρομερή σύγχυση γιατί αυτό που χρειάζονται οι παραγωγοί είναι μία καθαρή πορεία για το μέλλον. Αυτό λοιπόν το οποίο προτείνουμε τώρα είναι ένα γαλακτοκομικό ταμείο για να αναδομήσουμε τον τομέα. Και πράγματι, σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται αναδόμηση ο γαλακτοκομικός τομέας. Αν και νομίζω ότι υπάρχουν άλλες περιφέρειες όπου αυτή η πρόταση δεν είναι η ιδανική. Θα μου πείτε, αν δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο, από πού θα προέρθουν τα λεφτά Έχω την εντύπωση ότι αυτοί που προωθούν αυτή την πρόταση πιστεύουν ότι θα προέρθουν τα κονδύλια από τον πρώτο πυλώνα. Αλλά αυτό θα σημαίνει ότι θα, θα φτιάξουμε ένα κάστρο στον αέρα, χωρίς θεμέλια δηλαδή, ένα πύργο στην άμμο. Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2010 αφήνει ένα πάρα πολύ μικρό περιθώριο για τέτοιες ενέργειες και τα επόμενα χρόνια ο κίνδυνος ε, της... Ε, ε, ε, ε, δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι, είναι ορατός μπροστά στα μάτια μας και θα έχουμε πάρα πολύ λίγα χρήματα. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι μέσα στο κεφάλαιο 2, στον τίτλο 2, δεν υπάρχουν περιθώρια για ένα τέτοιο ταμείο. Αλλά βέβαια πρέπει να λάβουμε μέτρα και πρέπει να κάνουμε ορισμένα βήματα για την αναδόμηση. Αλλά όχι στα πλαίσια του τίτλου 2. Πιστεύω ότι αυτή η ιδέα του γαλακτοκομικού τομέα θα ήταν πολύ καλύτερη να είχε προταθεί το 2003. Αν τότε είχε ακουστεί αυτή η ιδέα που υπήρχε μία διάσπαση ε, των, του ανώτατου ορίου που μπορούσαν να λάβουν από ποσόστοση γάλακτος ή από την παρέμβαση. Ε, Παραδείγματο χάρη, οι Γερμανοί γαλακτοκοπαραγωγοί λάβαν τότε ένα δις ευρώ όχι μια, όχι μια φορά μόνο, αλλά κάθε χρόνο, όχι δηλαδή κατά αποκοπή, ε, αλλά μια, κάθε χρόνο ελάμβαναν αυτά τα χρήματα. Τώρα το, ο έλεγχος υγείας το, της ΚΑΠ, το CAP Health Check και το οικονομικό πρόγραμμα πακέτο ανασύστασης θα απελευθερώσει 4,2 δις ευρώ για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η αναδόμηση βεβαίως του γαλακτοκομικού τομέα. Αυτά είναι χειροπιαστά χρήματα, αληθινά χρήματα και πιστεύουμε ότι αυτά τα αληθινά, τα πραγματικά χρήματα χρειάζονται για την αναδιάρθρωση του τομέα και για να εξασφαλίσει το μακροπρόθεσμο μέλλον. Αυτή είναι η προτεραιότητα λοιπόν των ενεργειών μας και πιστεύουμε ότι αυτές οι ενέργειες μπορούν να, να ληφθούν, να γίνουν πραγματικότητα και να πραγματοποιηθούν μέσω των παραδοσιακών μέτρων ενίσχυσης ε, των αγορών και των ε, κρατικών ενισχύσεων μεταξύ άλλων ε, εργαλείων, μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και έτσι θα μπορέσουμε να ελέγξουμε και την κρίση της αγοράς. Το 2009 στον γαλακτοκομικό τομέα η επιπρόσθετο, το επιπρόσθετο κόστος για την επιστροφή εξαγωγών, αποπληρωμή χρεών κλπ, επιστροφή ποσών είναι 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά ε, τα χρήματα οφείλονται στην κρίση που έχει σημειωθεί και θα πρέπει να πληρωθούν μέσα σε 12 μήνες ε, το 12 μήνα δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2009. Αυτή τη στιγμή η κρίση αυτή η μεγάλη έχει ε, κάπως ομαλ... δείχνει σημάδια ομαλ... εξομάλυνσης και σταθεροποίησης και πιστεύω ότι τα ποσά αυτά ε, θα μειωθούν τα επόμενα χρόνια. Με την... Ε, για το 2009 και 2010 λοιπόν χρειάζονται περίπου ένα δις. Αυτά είναι τα ποσά τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να διαθέσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή που μας βοήθησε να λάβουμε αποφάσεις για τις, περίοδου για τις περιόδους ε, παρέμβασης του βούτυρο και στο αποκορυφωμένο γάλα υπό την απλουστευμένη διαδικασία και βασίζομαι στη συνεργασία σας για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά θέματα βούτυρο και αποκορυφωμένο γάλα. Όμως πιστεύω ότι η κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα είναι λάθος να την εξετάζουμε μόνο μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Σαφώς το βασικό πρόβλημα είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία έχει ε, την ζήτηση, τον τομέα της ζήτησης και δυστυχώ αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη τη δεν μπορεί να λύσει. Με ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα να δω τι γίνεται στη σχέση μεταξύ των γαλακτοπαραγωγών και της υπόλοιπης διατροφικής αλυσίδας. Οι τιμές παραγωγής για τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν πέσει κάτω από την, τις τιμές εχμής του 2007 όμως οι τιμές των καταναλωτή είναι ακόμα 14% υψηλότερες από ό,τι ήταν τότε, το 2007. Έτσι λοιπόν σκέφτομαι ότι η αλυσίδα διάθεσης και λιανικής πώληση έχει παίζει κάποιον ρόλο και δημιουργεί προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι στην αλυσίδα προμηθειών και διάθεσης υπάρχουν προβλήματα και θέλω να έχω ζητήσει από τους συνεργάτες μου να μου παρουσιάσουν μια αντελεχή ανάλυση των προβλημάτων και των ε, αντιφάσεων που υπάρχουν σε αυτήν την αλυσίδα. Επίσης, δεν πρέπει να χάνουμε τα μάτια μας, ε, το βλέμμα μας, από την ευρύτερη εικόνα που είναι η, η περαιτέρω ανάπτυξη του γαλακτοκομικού τομέα. Πρέπει να προσέχουμε πολύ σημαντικά πού πατάμε βραχυπρόθεσμα και πού στοχεύουμε μακροπρόθεσμα. Εάν χάσουμε αυτή τη μακροπρόθεσμη προοπτική θα χαθούμε τελείως σε έναν κικαιώνα. Έχει λοιπόν η ανάπτυξη της ΚΑΠ μετά το 2013 ξεκινήσει και με συζητήσεις λαμβάνουν μέρος και στο Συμβούλιο. Και υπάρχουν πάρα πολλέ ιστοσελίδες που αναφέρουν σε αυτό το θέμα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και όλες οι πτυχέ έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την παραγωγή, το περιβάλλον, την ε, ύπεθρο και την κοινωνία και, την κοινωνία και τις οικονομίες μας. Το γεγονός ότι η αγροτική παραγωγή βρίσκεται πάντοτε στις επικεφαλίδες και στις πρώτες σελίδες ε, του τύπου και των ειδήσεων δείχνει πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας και θα χρειαστούν τεράστιες προσπάθειες για να βρούμε τις σωστές απαντήσεις και τις οποίες δεν θα μπορέσουμε να βρούμε αν δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Πιστεύω ότι το φθινόπωρο του χρόνου, το καλοκαίρι το φθινόπωρο το αργότερο του χρόνου, η Κομισιόν θα μπορέσει να παρουσιάσει μια ανακοίνωση η οποία μεταξύ των άλλων θα προβάλλει και τις ιδέες της για την, με, για την εποχή μετά το 2013 και την ανάπτυξη της ΚΑΠ. Εν τω μεταξύ πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και εις βάθος συζητήσεις και βασίζουμε στη συνεργασία των μελών αυτής της Επιτροπής. Σήμερα το πρωί ε, διάλεξα να αναφερθώ σε τρία ακόμα συγκεκριμένα θέματα. Πρώτο, πρώτον, στις λιγότερο πλεονεκτικές περιοχές, τα less favored areas. Αυτό είναι άλλο θέμα το οποίο ε, για το οποίο συζητάμε με πολύ πάθος. Ε, πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι η Κομισιόν δεν έχει κάνει εδώ προτάσεις πολιτικής για αυτές τις λιγότερο πλεονεκτικές περιοχές. Ε, το 2005 άρχισε η συζήτηση να βρούμε έναν τρόπο αντικειμενικό να καθορίσουμε ποιες είναι αυτές οι μειονεκτικές, μειονεκτούσες περιοχές που έχουν τα φυσικά handicaps Πρέπει λοιπόν ε, να, ε, αν δεν έχουμε ένα σαφή ορισμό, υφιστάμεσα μία συνεχής επικρίσεις. Εάν λοιπόν δεν ολοκληρώσουμε αυτό το φάκελο, ε, θα είμαστε συνεχώς κατηγορούμενοι και θύματα μιας ε, ε, βάσιμης κριτικής. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ανακαθορίσουμε μια βασική ιδέα, μια κατευθυντήρια γραμμή για τις πληρωμές προς αυτές τις περιοχές, τις λιγότερο πλεονεκτικές περιοχές και γι' αυτό η Κομισιόν έχει παρουσιάσει τις αρχικές της ιδέες για 8 κριτήρια, καθορισμό 8 κριτηρίων που έχουν σχέση με το έδαφος, τις εδαφικές συνθήκες και το κλίμα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να κρίνουμε ποιες περιοχές έχουν ε, φυσικά εμπόδια ή μειονεκτήματα, τα natural handicaps και ποιες όχι. Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να περιλάβει ορεινές περιοχές ή περιοχές με συγκεκριμένα μειονεκτήματα αυτή είναι δηλαδή η ορολογία την οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά πριν παρουσιάσουμε ένα, μία πρόταση με νομική βάση, θα ήθελα να δω αν το σύστημα θα, θα δουλέψει πρακτικά. Γι' αυτό λοιπόν έχω καθορίσει μία προθεσμία μέσα στα οποία τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν του χάρτε στου οποίου θα δείχνουν αυτέ τι περιοχέ και πού θα εφαρμοστούν αυτά τα κριτήρια μέχρι τον Ιανουάριο του 2010. Προφανώς λοιπόν καταρχάς πρέπει να καθορίσουμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές, οι, τα LFAs και εν συνεχεία να κάτσουμε και να ανασκουμποθούμε και να δουλέψουμε για να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα κριτήρια. Είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε τα ε, κριτήρια τα οποία θα μας κατευθύνουν στις μελλοντικέ αποφάσεις. Ε, πολύ πιο σημαντικά από την μείωση των πληρωμών ή περιορισμό των περιοχών αυτών, εκτάσεων αυτών. και δεν θα ήθελα το θέμα αυτό να, να επισκιαστεί από τα σημερινά παγκόσμια προβλήματα της οικονομίας. Βεβαίως ε, οι άνθρωποι μέσα στο, στον κικαιόν αυτής της κρίσης ε, αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες ή αλλάζουν ε, ορισμένες τον τρόπο με τον οποίο τρώνε ή τα φαγητά που διαλέγουν ή αγοράζουν αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς πρέπει να παραμείνουμε ισχυροί παίκτες στην ε, παγκόσμια αγορά και θα πρέπει να παραμείνουμε, ε, θα πρέπει να, ε, να είναι εμφανής ο ηγετικός μας ρόλος στην αγροτική πολιτική ποιότητος. Επίσης, προχωρούν οι εργασίες μας ε, για, μέσα στα πλαίσια της, ε, του αγροτικού τομέα για, ε, στην αλλαγή του κλίματος που αποτελεί μια προτεραιότητα της Σουηδικής Προεδρίας και πιστεύω είναι η παρισμόν ένα πρόκληση του μέλλοντος θα επηρεάσει λοιπόν ε, σημαντικότατα η, πολιτική της αλλαγής ε, του κλίματος ε, την παραγωγή, την αγροτική παραγωγή διότι πρέπει σαφώς να μειωθούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και έτσι έχουμε από τη μία πλευρά να εξασφαλίσουμε την επάρκεια προϊόντων τροφίμων την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος. Μια πολύ δύσκολη ισορροπία πρέπει να βρεθεί εδώ, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Η ΚΑΠ ε, διαθέτει πολλά μέσα, πολλά, πολλές πολιτικές που μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε πάνω σε αυτή ε, την προοπτική ε, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος μετά το 2013. Επίσης ε, θα προσέλθουμε με, με μεγάλο δυναμισμό στις συζητήσεις ε, που θα γίνουν το Δεκέμβριο στην Κοπενχάγη στη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ ε, για την αλλαγή του κλίματος. Θα, θα ακούσω τις ερωτήσεις σας βεβαίως πολύ σύντομα αλλά θα ήθελα να καταλήξω με ορισμένα σχόλια ακόμα το, πρέπει να πω ότι το κοινοβούλιο, αυτό, αυτό το, το έτος το κοινοβούλιο θα ε, έχει μια, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που θα έχει μια μεγάλη επίπτωση στην καλή μας συνεργασία. Και αυτό το σημαντικότερο το γεγονός που θα συμβεί είναι η αλλαγή ε, των αποφάσεων για την ε, ΚΑΠ. που θα πλέον ενταχθούν στο πλαίσιο της συναπόφασης. Βέβαια, θα πρέπει να μάθουμε, να, να, να κάτσουμε σαν μαθητές και να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα, αλλά πρέπει να σας μεταδώσω ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την Κομισιόν ε, προς την Επιτροπή σας. Είμαι πολύ, πολύ ικανοποιημένη ότι η ΚΑΠ θα περιέλθει στην αρχή της συναπόφασης ε, και το Κοινοβούλιο θα είναι ισότιμος εταίρος με το Συμβούλιο διότι έτσι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε καλύτερα τις σχέσεις μας που θα βασίζεται στην απόλυτη εμπιστοσύνη ε, στην πλήρη συνεργασία και ισότιμη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και ξέρω ότι και ο Πρόεδρος θα συνεργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς ε, βεβαίως η συναπόφαση απαιτεί ε, περισσότερο χρόνο για να εξετάζουμε μαζί τις νομοθετικές πτυχές. Αλλά είμαι βέβαιη ότι αυτό το πλαίσιο συναπόφασης θα προσδώσει ακόμα περισσότερη νομιμότητα στις αποφάσεις μας. Η καλή νομοθεσία βασίζεται εν μέρη στη γνώση, στο θησαυρό των γνώσεων και όπως σε, πολλές, σε πολλούς άλλους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής, η ΚΑΠ, δεν είναι ένα κεφάλαιο το οποίο μπορεί κανείς να το περάσει στο γόνατο και να τα μάθει όλα ε, με ένα φάκελο στα γόνατά του καθήμενος μπροστά στην τηλεόραση το ξέρω αυτό και ξέρω ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή γνώσεων στην Επιτροπή σας και εγώ θα βοηθήσω όσο μπορεί περισσότερο να αναπτύξουμε αυτή τη δεξαμενή γνώσεων. Ο πρόεδρος Ντεκάστρο μας ζήτησε ε, να διοργανώσουμε μια σειρά τεχνικών briefings και βεβαίως η Κομισιόν, ενημερώσεων δηλαδή, και βεβαίως η Κομισιόν θα κάνει αυτές τις ενημερώσεις, αυτά τα briefings. Η η ενδελεχή συζήτηση, ε, η συμμετοχή σας με πάθος και αποφασιστικότητα, αυτά είναι τα, τα, μεγάλα πλεονεκτήματα της Επιτροπής σας. Και είμαι βεβαία ότι δεν θα με αποκοητεύσετε. Θα συνεργαστούμε με τον ίδιο δυναμικό και αποφασισμένο τρόπο και στο μέλλον σε αυτό το φθινόπορο που μας έρχεται. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Μαρία για αυτή την παρουσίαση που μας έκανες ε, σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην συζήτηση. Πάρα πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Προς το παρόν έχουμε 22 εγγεγραμμένους. Εγώ φυσικά είμαι υποχρεωμένο ε, να τηρήσω κάποια χρονικά περιθώρια για να επιτρέψω σε όλους σας να λάβει το λόγο. Υπενθυμίζω πως είχαμε μια μακρά συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι κατανοήσαμε πως ε, απαιτείται να δράσουμε περαιτέρω στον γαλακτοκομικό τομέα. Προς το πάνω θα δώσω το λόγο στους συντονιστές ε, χρόνο δύο λεπτών. Κάθε συντονιστή λοιπόν έχει δύο λεπτά στη διάθεσή του και μετά θα ακολουθήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δυστυχώ για ένα μόνο λεπτό για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τι εργασίε των 12 και 30. Ξεκινάμε με τον Αλμπερτέ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήρθατε ακριβώς στην αρχή της ε, νέας ε, περίοδου εργασιών μας. Είχα μεγάλες επιφυλάξεις ε, για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής και της καταστάσεως των παραγωγών μας. Βλέπω πολλούς επαγγελματίες συναδέλφους που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα με τις τιμές του γάλακτος έχουμε μία τέτοια μείωση, μία τέτοια φθορά που ε, ακόμα και οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες δεν θα μπορέσουν πολύ σύντομα να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή το κόστος παραγωγής έχει θα ξεπεράσει, αν δεν έχει ήδη ξεπεράσει την τιμή του γάλακτος, ε, την τιμή διάθεσης. Οπότε υπάρχει μεγάλη πικρία μεταξύ των παραγωγών, ιδίως αυτών που λαμβάνουν το κατώτερο επίπεδο πληρωμής. Όπως ξέρετε, αυτή η κατάσταση έχει και μια κακή ψυχολογική επίπτωση το εμπόριο, ο εμπορικός τομέας έχει πάρα πολύ σημαντικά μειώσει τις τιμές. Και στις 12 Μαρτίου του περασμένου έτους είχα πει ότι μετά από αυτή την απόφαση μειώσεως των τιμών και είχα πει κυρία Επίτροπε ότι αυτή η, η, η διεύρυνση των ποσοστώσεων δεν θα οδηγήσει σε μια ομαλή προσγείωση με το νέο καθεστώς δηλαδή του μέλλοντος αλλά θα οδηγήσει σε συντριβή σε συντριβή των παραγωγών. 7, 8, 7, 8 ευρώ ανά 100 κιλά ε, δημητριακών δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτού του τομέα. Γι' αυτό είχα προτείνει μέχρι είχα πει μάλλον ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου θα δούμε τεράστιες χρεοκοπίες και συντριβή μεγάλων παραγωγικών μονάδων λόγω της καταστάσεως των τιμών. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη αυτή την πάρα πολύ δυσμενή κατάσταση του τομέα. Σας ευχαριστώ κύριος Κάπολα Σάντος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα... να υπενθυμίσω και να ονομάς της ομάδας μου πως είμαστε απόλυτα διατεθειμένοι να συνεχίσουμε μια ειλικρινή και έντιμη συνεργασία όπως εξάλλου είχαμε και κατά την προηγούμενη θητεία μας. Κυρία Επίτροπε θα είμαι σύντομος. είπατε κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά δεν με ευχαρίστησαν διόλου. Όντως η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στον γαλακτοκομικό τομέα και δεν είναι η στιγμή να ξεκινήσουμε κάποιες ε, δογματικές ή ιδεολογικές συζητήσεις. Είμαι φιλελεύθερος, ε, ε, σέβομαι τις απόψεις αλλά έχω και εγώ δικές μου. Κρίνω πως η σημερινή κατάσταση απαιτεί λύσεις πραγματιστικές και Σοβαρέ. Δεν γνωρίζουμε πώ έχει κατάσταση. Ως πολιτικοί θα πρέπει να διασφαλίσουμε την σταθεροποίηση των αγορών αλλά και λογικές τιμέ τόσο προς τους παραγωγούς όσο και προς τον καταναλωτή. Ως ε, πολιτικοί εκπρόσωποι νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε στο ύψο των περιστάσεων. Είπατε ότι η αγορά θα τίνει σε μια κατάσταση σταθερότητα, αλλά αυτό δεν ε, οδηγεί και σε επιβίωση του κλάδου. Εμείς δεν θέλουμε σταθερότητα, μπορεί να θέλουμε σταθερότητα μένα, αλλά θα πρέπει να εγγυηθούμε στους παραγωγούς την επιβίωσή τους. Και πάρα πολλοί γεωργοί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ε, με τις τιμές που ισχύουν δεν μπορούν να επιβιώσουν. Είναι μια έκτακτη κατάσταση η οποία απαιτεί έκτακτα μέτρα. Είμαι απογοητευμένος διότι ήλπιζα πως ε, πριν από ε, ένα συμβούλιο υπουργών το οποίο θα συνέλθει εκτάκτως και μην ξεχνάμε ότι συνήλθε στις 27 του μήνα το, η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε μάλλον και ελπίζαμε κυρία Επίτροπε ότι θα μας υποβάλλετε προτάσεις εντάξει η Κομισιόν έδειξε καλή βούληση αλλά είμαστε πεπισμένοι πως τα μέτρα είναι ανεπαρκή πρέπει λοιπόν να πάμε παραπέρα τόσο ε, εγώ όσο και οι συναδελφοί μου υποβάλαμε κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού θα πρέπει για μια περιορισμένη περίοδο να ε, δράσουμε ασκώντας πίεση στις αγορές. Υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης των δημοσίων αρχών. Ας μην αφήσουμε λοιπόν την αγορά στα χέρια των ε, της ελεύθερης οικονομίας. Ε, διαφορετικά θα οδηγήσουμε την, ε, τους ε, γεωργούς σε χρεοκοπία. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την σωστή λειτουργία της αγοράς, οποιαδήποτε και αν είναι τα μέτρα που θα απαιτηθεί να λάβουμε. Θέλαμε λοιπόν να πάρετε ξανά το λόγο και να μας πείτε τι, τι ποια είναι η απόψη σας για αυτή την κατάσταση. Τα λόγια σας πραγματικά δεν με καθησύχησαν. Εντάξει, δείξατε πολύ καλή βούληση και ευχαριστώ τον πρόεδρο που μου έδωσε το λόγο. Το λόγο έχει ο Τζιμ Νίκολσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σας βλέπω πάλι ανάμεσά μας. Είπατε πως ε, η κατάσταση είναι σοβαρή, όλοι το γνωρίζουμε, οι Γεωργοί δεν είχαν ποτέ αντιμετωπίσει τόσο σκληρές συνθήκες ε, και να χρειάζονται να παράγουν κάτω του κόστους, ε, να πολλούν συγγνώμη κάτω του κόστους. Εμεί δεν θέλουμε να δώσουμε μια βραχυπρόθεσμη απάντηση στο πρόβλημα. Πρέπει να εξεύρουμε μια λύση μακροπρόθεσμη, μακρόπνοη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δουλέψουμε χέρι-χέρι και να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ε, το τι θα συμβεί μετά το 2015 είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε προσοχή, αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να ε, λύσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γαλακτοπαραγωγή. Χρειάζεται λοιπόν να τους ενισχύσουμε. Αυτό το γνωρίζω από την δική μου περιοχή, αυτό το γνωρίζω πίσω ότι σημαίνει και σε άλλες περιοχές. Ένας από τους ε, τομείς λοιπόν που μας προβληματίζει είναι η διαφορά την οποία του τιμή που λαμβάνει ο παραγωγό και η τιμή του που έχουμε στα καταστήματα του σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει λοιπόν να ασκηθεί κάποιο έλεγχο. Εδώ έγκυται λοιπόν το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να υποχρεώσουμε του ε, μεγάλε αλυσίδε να καταβάλουν ένα σωστό, μια σωστή τιμή στους ε, παραγωγούς και κάτι ακόμα. κάτι το οποίο είδαμε κατά τη διάρκεια του θέρους το θέμα της ε, έγκρισης Αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο μας προβληματίζει. Διερωτώ λοιπόν κατά πόσο η σημερινή συζήτηση το απόγευμα θα μπορέσει να βοηθήσει και στην επίλυση του θέματος που αφορά στο, στην εισαγωγή βραζιλιανικού κρέατος. Μάρτιν Χόσλιν έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, και εκ μέρους των Πρασίνων εύχομαι μια καλή συνεργασία και σας προσφέρω την καλή συνεργασία από το, την ομάδα μας. Ήλπιζα οι καλοκαιρινέ διακοπές να σας είχαν εμπνεύσει και να μας είχατε έρθει με καινούργιε ιδέες. Αλλά αυτό που βλέπω είναι μία από τα ίδια από αυτά που άκουσα. Ε, ένα χαμηλό επίπεδο δηλαδή προτείνεται, το οποίο σαφώς δεν θα εγγυηθεί το εισόδημα, το γαλακτοπαραγωγό στο μέλλον. Όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία, τα μέτρα τα οποία αναφέρατε είναι 600 εκατομμύρια ενίσχυση εξαγωγών και δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστός τρόπο να ξοδεύετε 600 εκατομμύρια για εξαγωγές για να φέρετε μια ισορροπία στην αγορά ενώ θα έπρεπε να επέλθει η ισορροπία στο όλο καθεστώ των ε, ποσοστώσεων οι οποίες θα καθαργηθούν έτσι κι αλλιώς μετά το 2015 αλλά μέχρι τότε πρέπει να δουλέψουμε με τις ποσοστώσεις Άρα λοιπόν η σωστή κατεύθυνση είναι να μειωθούν οι ποσοστώσεις. Αυτό θα δώσει το σωστό μήνυμα στην αγορά. Εδώ το πρόβλημα είναι ε, τα ποσά ε, και όχι η ζήτηση. Ε, δυστυχώς λοιπόν δεν σας ενέπνευσε το καλοκαίρι και δεν βλέπω πώς με αυτά που είπατε θα βρεθούν λύσεις. Κάθε μέρα χάνονται θέσεις εργασίας, κάθε μέρα μειώνεται ο τομέας κάθε μέρα στις λιγότερο στις μειονεκτικές περιοχές της ε, ε, μη μειώνονται οι παραγωγικές μονάδες και γι' αυτό είναι επίγουσα η δράση την οποία πρέπει να αναλάβουμε. Ε, πιστεύω ότι πρέπει, αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβουμε μέτρα άμεσα γιατί οι επιπτώσεις είναι ε, πολύ αρνητικές. Τώρα, για την ενίσχυση των εξαγωγών και αυτά τα, το ποσό που θέλετε να διαθέσετε, δεν είναι λύση. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται μία φθήνουσα πορεία διεθνώς στο, στην παγκόσμια αγορά ενίσχυση των εξαγωγών ε, δεν είναι, θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα σε ορισμένες ε, χώρες. Δεν είναι λοιπόν μία λύση γενικός γενικώ για όλους η ενίσχυση των εξαγωγών και ε, πιστεύω ότι η ανισορροπία στις αγορές γάλακτος θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το καυτό πρόβλημα των ποσοστώσεων και της μελλοντική τους κατάργησης. Ένα Άλλο θέμα που με ενδιαφέρει είναι τι θέματα θα τεθούν ε, στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων στην Κοπεχάκη. Η ατζέντα δηλαδή και τα συγκεκριμένα θέματα, τι θα προτείνετε εσείς. Και εν συνεχεία το, τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα στις εισαγωγές και στις αγορές τροποποιημένων προϊόντων. Η Μέρι Πόλσον. Μέρι Πόλσον, παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο σας, λέει ο Πρόεδρος. Είμαστε πιεσμένοι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε. Δεν θέλω, δεν έχω να πω τόσα πολλά για αυτήν την ε, μεγάλη κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα. Πρέπει οπωσδήποτε η προοπτική μας να είναι μακροπρόθεσμη, μια συνολική προοπτική να εξετάσουμε για τα μέτρα μας όπως και οι πράσινη πιστεύω και εγώ ότι η ενίσχυση των εξαγωγών θα οδηγήσει σε μια ακόμα πιο ε, φθήνουσα και κατηφορική πορεία, ένα σπυρά δηλαδή προς τα κάτω. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, μεγάλη κρίση αυτή με άμεσα μέτρα ενίσχυσης. Δηλαδή, κάτι το οποίο δεν θα είναι μόνιμο, δηλαδή τα ε, μέτρα ενίσχυσης δεν θα είναι μόνιμα, δεν θα παγιωθούν, αλλά θα, θα εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστεί η έκτακτη αυτή τεράστια κρίση. Η γαλακτοπαραγωγή, όλοι οι στον τομέα, είναι αυτοί που υποφέρουν με τις τιμές που λαμβάνουν σε σχέση με τις τιμές πώλησης στο λιανικό εμπόριο. Πρέπει λοιπόν σαφώς να εξετάσουμε τι συμβαίνει μεταξύ της τιμής που δίνεται στο γαλακτοπαραγωγό και της τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής για να αγοράσει το γάλα του και τα συναφή προϊόντα. Αυτή η αλυσίδα λοιπόν πρέπει να αναλυθεί και να ε, εντοπιστούν τα προβλήματα. Και το γρηγορότερο μάλιστα το φθινόπωρο αυτό θα πρέπει να αποφασίσουμε για μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν το μέλλον του τομέα. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε κοντόφθαλμα να ξεπεράσουμε ποτέ αυτή την κρίση η οποία έχει δημιουργήσει εκατομμύρια ανέργους στην Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα από μέτρα, από ε, άμεση ενίσχυση των παραγωγών. Εάν θέλουμε να αναπτύξουμε την Ήπεθρο και αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ποικιλομορφία της υπαίθρου, τις πολιτιστικές ε, πτυχές και τη ζωή στην υπαίθρο θα πρέπει να χειριστούμε αυτά τα προβλήματα διαφορετικά θα υποφέρουμε. Το λόγο έχει ο Αλφέντ Ρούμπιξ ε, ως τελευταίος ομιλής από πλευρά της επικεφαλής ομάδα. Τα θέματα αυτά που άπτονται της γεωργίας και κυρίως τα γαλακτοκομικά ε, προβλήματα ε, είναι, πολύ, είναι ζωτική σημασία για τη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ένα μέρος της ευθύνης για την κρίση που αντιμετωπίζουμε στην χώρα μου. Και η κρίση δεν αφορά μόνο τον γεωργικό τομέα ή τον γαλακτοκομικό τομέα, είναι γενικότερη. έχουμε δανειστεί, το, έχουμε δανειστεί 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το, το μισό τουλάχιστον από το ΑΕΠ μας και οι, οι γεωργοί μας προσπαθούν να πουλήσουν απεγνωσμένα τα προϊόντα τους συναντούν όμως όλο ένα και περισσότερες δυσκολίες. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους ότι τα μέτρα τα οποία προτείνονται αυτή τη στιγμή για να σταθεροποιηθεί ο γεωργικός τομέας είναι αναξιόπιστα και ανεπαρκή. Εάν αποτύχουμε την διατήρηση μιας υγιούς γεωργίας δεν θα έχουμε πετύχει έναν από τους βασικούς μας στόχους που είναι δηλαδή να εξασφαλίσουμε την αυτάρκεια στα γεωργικά προϊόντα. Και υποστηρίζω την ε, συνέχιση της ε, συζήτησης αυτής, διότι θα πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, διαφορές ε, στο τι μπορεί να πετύχουν τα μεγάλα και τα μικρότερα κράτη-μέλη. Κυρίως ε, στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις 25 συναδέλφων που έχουν ε, εγγραφεί και στις 12 και 4 πρέπει να δώσω και τον λόγο στην Επίτροπο για να απαντήσει. Ε, εάν ε, είμαστε... αν ακολουθήσουμε την, μια πειθαρχία θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Αλλιώς οι τελευταίοι δεν θα μιλήσουν. Α, 30 δευτερόλεπτα. Ε, άντε ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επιτροπέ. Θα μιλήσω για, την, για τα γαλακτοκομικά και την κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα. Είναι γενικότερη κρίση. Ε, και εσείς πέρυσι είσαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Μας ήρθατε ξαφνικά. Πώς θα διαχειριστούμε όμως αυτή την κρίση που είναι πρόβλημα προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση. Έχουμε πάρα πολύ γάλα, βάζουμε ε, σε ενέργεια διάφορα μέτρα, παρέμβαση, στήριξη κτλ. κτλ. Και υπάρχουν δύο διαρθρωτικοί δρόμοι για να λύσουμε την κρίση. Αυτή την οποία προτείνεται και την οποία δεν μπορώ να αντιδεχτώ, δηλαδή η διάρθρωση μειώνοντα τον αριθμό των παραγωγών. Ένα αυτό, ένα σενάριο αυτό. Δεύτερον, να επανέλθουμε ε, και να αλλάξουμε τις αποφάσεις που έχουμε πάρει που είναι αντιφατικές σε σχέση με αυτά τα οποία εστίνουν τώρα. Λοιπόν τώρα που δίνουμε επιδοτήσεις και παρέμβαση από τη μια πώς αυξάνουμε τις ποσοστώσεις κατά 1% ε, τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να επανέλθουμε στην απόφαση αυτή. Ένα αυτό. Δεύτερον, αν πρέπει να δοθούν βοήθειες και ενισχύσεις, θα πρέπει να δίδονται κυρίως στην, ε, να είναι μέτρα υποστήριξης του εισοδήματος και όχι να χρηματοδότηση τη διάρθρωση των διαρθρωτικών μέτρων που θα οδηγήσουν σε μείωση των, του αριθμού των παραγωγών του, κατά κάτω δεν φταίνει η παραγωγή για την ε, κατάσταση αυτή. Ε, άλλο θέμα. Εάν αν καταργήσετε τι γαλακτοκομικέ ποσοστώσεις, τι θα εφαρμόσετε στη θέση αυτών, όταν γνωρίζουμε ήδη ότι πολλέ φορέ ε, τι ποσοστώσεις ε, τις ξεπερνάνε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Αυτά είναι, αυτά είναι τα ερωτήματα που σα θέτω και τα προτάσεις οποίες κάνω. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη μου παρέμβαση και θα ήθελα να χαιρετήσω την Επίτροπο αλλά και όλου τους συναδέλφους. Αναφέρθηκαν δύο θέματα μεταξύ των άλλων. Πρώτα απ' όλα η ποιότητα των προϊόντων και τα ε, φυσικά ελλείμματα ε, που υπάρχουν. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το θέμα έχει μεγάλη σημασία για τις Κανάριες νήσους ε, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο ζήτημα της ε, μπανάνας. Ξέρουμε ότι ο πόλεμος της μπανάνας υπήρξε και θα συνεχίσει να υπάρξει. Εμένα μένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το μέλλον των Ευρωπαίων παραγωγών της μπανάνας. Ξέρουμε λοιπόν ότι ε, χρειάζεται να τους χορηγηθεί κάποια βοήθεια. Και αυτό αφορά επίσης και τους ε, εταίρους μας της Λατινικής Αμερικής. Θα ήθελα να σας ζητήσω ε, να αποτελέσει προτεραιότητα για την Κομισιόν η προστασία των παραγωγών της μπανάνας. Και να πω κάτι ακόμα για την ντομάτα. Και εδώ θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς και την περίπτωση των Καναρίων Ίσων αυτό απαιτεί μια συμφωνία αλλά και για ολόκληρη την Ισπανία θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να τηρηθούν τα συμπεφωνημένα και ειδικά σε ό,τι φορά συμφωνείς με το Μαρόκο. Οι απαιτήσει λοιπόν της ε, Ευρώπης θα πρέπει να ισχύουν και για τις υπόλοιπες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπη, είχα ένα διάλειμμα δύο ετών πριν ξανάρθω εδώ. Ε, και χαίρομαι που γυρίσα πίσω μεν, αλλά αντιμετωπίζουμε μια κρίση μίζωνος σημασίας. Το πρόβλημα ποιο είναι. Αυτή η το, η αγορά η οποία αλλάζει συνέχεια. Είτε είναι το σιτάρι, είτε είναι ε, το γάλα τώρα, ε, αυτές οι αλλαγές που γίνονται, οι συνεχείς αλλαγές ε, δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Όντως δεν πρέπει να δράσουμε μέσω μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα κυρίως. Όμως αν δεν δράσουμε και βραχυπρόθεσμα θα εξαφανιστούν ε, χιλιάδες γεωργοί. αναφέρθηκαμε και στις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις. Η, αυτή την πρόταση που μας κάνετε δεν μπορούμε να τη δεχτούμε για την διάρκεια η ρύθμιση όμως που είπατε, εσεί αναφερθήκατε στη ρύθμιση, είπατε ότι η αγορά θα πρέπει να φτάσει σε μια ε, ισορροπημένη κατάσταση. Ποια θα είναι αυτή η ισορροπία όμως, ε, πρέπει να είναι μια ε, ε, σοβαρή ισορροπία και έντιμη ισορροπία. θα πρέπει να μιλάμε για μια λογική τιμή και θα πρέπει να σεβαστούμε και την ποιότητα. Λοιπόν, θα, θα, εσείς πώς το βλέπετε αυτό να έχουμε μια λογική τιμή εξα, ε, εξασφαλίζοντας και την ποιότητα και αυτό να οδηγεί σε μια ισορροπία των αγορών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και την Επίτροπο. Μια και έχω ένα λεπτό, τρία λεπτά για το γάλα. Αναφερθήκατε ότι, είστε, ότι οι παραγωγοί θέλουν να ξέρουν τι πρόκειται να συμβαίνει, να συμβεί στο μέλλον. και συμφωνώ μαζί σας, όμως θα πρέπει να ε, θέσουμε το ερώτημα ως εξής, όπως είπε και ο συνάδελφος. Με τι θα αντικαταστήσουμε το ποσοστό, τις ποσοστώσεις και οι γαλακτοπαραγωγοί θα ακολουθήσουν τους παραγωγούς των Δημητριακών, δεν θα έχουν καμία υποστήριξη. Ε, δηλαδή, εάν είναι αν τελείως ελεύθερη η παραγωγή, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την αγορά. Διότι, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, η κατάσταση δεν είναι απλώς μόνο σοβαρή, είναι ε, είναι στο χειρότερο, ε, στην χειρότερη κατάσταση που μπορούμε να φανταστούμε, διότι ε, κινδυνεύουν τα εισοδήματα των γεωργών, κινδυνεύουν με οι γεωργοί και οι οικογένειές τους να χάσουν τελείως τα εισοδήματά τους. Και ε, κάτι χρειάζεται, χρειάζεται να γίνει. Ε, ακούω για τους μεταποιητές να λένε κάτι για το τυρί, δεν κάνουμε όμως σοβαρά πράγματα. Ε, επίσης, για την εισαγωγή πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα δημιουργηθεί μια κρίση. Άκουσα διάφορα φήμες και απόψεις που αφορούν και το θέμα των μεταλλαγμένων. Αλλά εσείς μπορείτε να Μα πείτε κάτι για, την, για τις προμήθειες σε πρωτεΐνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Παπαστάμπος Κύριε Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο για την ανάλυση της. Ως μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, στην προηγούμενη θητεία υπήρξα εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις του γύρου της Δόχα στο Χονγκ Κονγκ, αλλά και έλαβα μέρος σε επισκέψεις, συναντήσεις με τους αρμοδίους του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου στη Γενέβη. Τότε υπήρξε το διαπραγματευτικό offer, η διαπραγματική προσφορά το Οκτωβρίο του 2005, η οποία ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη, δεν βρήκε ανταπόκριση από άλλους εμπορικούς μας εταίρους, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να παραχωρήσει χωρίς να υπάρχει η αρχή της αμοιβαιότητας, χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση από άλλους κορυφαίους εμπορικούς δεόντες στον κόσμο. Αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις του γύρου της Δόχα εκ νέου, μετά την αποτυχία του Ιουλίου του 2008. Θα υπεραμεινθείτε, κυρία Επίτροπε, των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Γεωργίας ή θα αφήσετε την Επίτροπο Διεθνούς Εμπορίου να βάλει τη σφραγίδα στη διαπραγματευτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συνεχίσετε στη γραμμή που τηρήσατε και το 2005. Υπάρχει εκείνο το offer ε, υπάρχει εκείνο το mandate, υπάρχει εκείνο το mandat, τι πρόκειται να γίνει από πλευράς ε, Κομισιόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για, την, ε, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Δεν είμαι προστατευτικός, αλλά θέλουμε ένα πραγματικά δίκαιο εμπόριο, ένα fair trade και όχι άλλες αντιλήψεις τελείως νεοφιλελεύθερες που πάνε να επικρατήσουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Państwa, w κατά τη γνώμη μου, απαιτεί να έχουμε πάντα υπόψη μα το μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Η ερώτηση είναι μήπως η σημερινή κρίση οφείλεται σε λάθη που κάναμε στο παρελθόν. Άρα λοιπόν πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη για την μελλοντική μα στρατηγική. Η σημερινή κατάσταση οφείλεται και εν μέρη στην ε, πολύ μικρή ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι μόνο το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της μείωσης της ζήτησης. Αναρωτιέμαι τι μπορεί και τι θέλει να κάνει η Κομισιόν για να ξεπεράσει αυτή τη μεγάλη διακύμαση των τιμών που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Έχετε αναλύσει τα αίτια των διακοιμάσεων των τιμών, γιατί προέρχονται και από πού. Και η επόμενη ερώτηση. Έχουν συναχθεί ε, συμπεράσματα από τη μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης. Ποια είναι τα συμπεράσματα αυτά, τι είναι τα μαθήματα τα οποία λάβαμε από αυτή τη μεταρρύθμιση. Επίσης, άλλη ερώτηση που αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ε, τι συζητήσεις θα, σε τι συζητήσεις θα συμμετάσχετε και τι θέματα θα προβάλλετε στα πλαίσια του ΠΟΕ. Και άλλη μια ερώτηση, τι πιστεύετε ότι, ε, ποιες θα είναι οι προβλέψεις του μέλλοντος για τον ε, πληθυσμό της γης, της υφηλίου και τι προγραμματισμό θα πρέπει να κάνουμε για παραγωγή, για την αγροτική παραγωγή ανάλογα με την πληθυσμιακή αύξηση σε συγκεκριμένα μέρη του πλανήτη. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελόγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πίτροπο που βρίσκεται πάλι εδώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τη βλέπουμε και που είναι μαζί μας θα ήθελα να προσθέσω ακόμα κάτι σε σχέση με τον τομέα του γάλακτος. Θα ήθελα να είχα ακούσει πιο φιλόδοξους στόχους για την ενίσχυση του τομέα. Και επίσης ε, δεν αναφέρεται την ανταγωνιστική θέση του τομέα αυτού και ακριβώς τι εύρος θα έχουν οι κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την ανάλυση της αλυσίδας ε, της παραγωγής ε, τροφίμων και ιδίω το γάλα, τι μεγάλε διαφορέ από την τιμή παραγωγή στην τιμή πώληση, χαίρομαι ιδιαίτερα που θα αναλάβετε μια τέτοια ανάλυση. Δεν θα πρέπει όμω ταυτόχρονα να εξετάσετε και τον ανταγωνισμό και να δείτε σε ποιες περιοχές του κόσμου οι παραγωγοί έχουν οργανωθεί καλύτερα και έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Ε, βεβαίως εμείς βλέπουμε πάντοτε από τη σκοπιά των, Βρυξελών. Αλλά εάν θέλουμε να αποζημιώνουμε σωστά τους, τους παραγωγούς υπάρχει και το θέμα των συγχωνεύσεων. Μήπως θα πρέπει να προωθήσουμε και αυτή την ιδέα. Και όσον αφορά την αποζημίωση ε, για θέματα περιβάλλοντος, αυτή μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Από τη μία κρατική ενίσχυση, από την άλλη αποζημιώσεις για το περιβάλλον, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Äh, Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα ε, στην ε, ειδική θέση και στα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν η παραγωγή στην Ήπεθρο και ε, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές. Η κρίση έχει επηρεάσει ιδιαίτερα του γαλακτοπαραγωγού στι ορεινέ περιοχέ, όπου δεν υπάρχει και μεγάλη προοπτική τουριστική ανάπτυξη και σε απομακρυσμένε ορεινέ περιοχέ, υπάρχουν ορισμένε περιφέρειε ορεινέ που σα έχουν υποβάλει συγκεκριμένε προτάσει στα πλαίσια τη ΚΑΠ για την ανάπτυξη συγκεκριμένης, περιοχής, ε, συγκεκριμένης πολιτικής ενίσχυσης των απομακρυσμένων ορεινών περιοχών. Παρακαλώ, λάβετε υπόψη αυτές τις προτάσεις που τις έχετε ήδη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω κυρία την, κυρία Επίτροπο και εγώ είμαι παλιός φίλος από την προηγούμενη θητεία, όχι τόσο παλιός όσο άλλοι συνάδελφοι τέλος πάντων. Εγώ είμαι από τη Σκωτία και ήθελα να πω ότι ε, αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με τα γαλακτοκομικά προϊόντα και με τις ποσοστώσεις ε, και αντιμετωπίζουμε προβλήματα διότι άλλες χώρε δεν έχουν σεβαστεί τι ποσοστώσεις αυτές και φοβούμε ότι ε, οποιαδήποτε Οπότε κριτήρια εφαρμόσουμε θα είναι, θα είναι περιτά λόγω της αν, ανυπαρξίας ή της μη επάρκειας του, του γεωργικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού για τις ποσοστώσεις. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Γκαρσία Περέθ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συμφωνώ το... με τα όσα είπατε σχετικά με το ότι υπάρχει διάλογος και συνεργασία μεταξύ ημών και ημών. Τώρα σχέση με την κρίση στον ολοκληρωτικό τομέα συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων σχέση με τα όσα έγιναν με την ανακοίνωση των Κομισιόν. Εσείς μιλήσατε για ενίσχυση. Δεν με ακούτε κύριε Επίτροπε. Υπάρχει πρόβλημα. μας ε, μιλήσατε για τον γαλακτικό τομέα και για την κρίση και ότι εσείς ζητάτε να εμβαθυνθούν περαιτέρω τα μέτρα. Αλλά όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή κρίση χρειάζονται να ληφθούν ευρωπαϊκά μέτρα. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε μόνο στα χέρια των κρατών μελών και των ενισχύσεων, αλλά να προωθηθούν κοινοτικά μέτρα τα οποία θα αντιμετωπίσουν τον στο οικονομικό τομέα. Και να κάνω μια ερώτηση γενικότερου χαρακτήρα σχετικά με τις τιμές. Τι πρόκειται να πράξει η Κομισιόν προκειμένου να βελτιωθεί η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις ε, τιμές καρναλωτή και τιμές παραγωγού. Ε, ε, πρόκειται για κάτι το οποίο επανειλημμένα έχουν αναφέρει οι παραγωγοί ιδιαίτερα στη χώρα μου. Υπάρχουν διαφορές όπως το γιόμιλο Τη τάξη του 1100 ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και την τιμή καταναλωτή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα προωθήσει η Κομισιόν σχετικά με τέτοια ζητήματα. Ευχαριστώ. Ζωζέ Μποβέ. Καλημέρα κυρία Επίτροπε. Γνωριζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια και συναντηθήκαμε και στις διαπραγματεύσεις για τον ΠΟΕ. Ήθελα να σας πω ότι σήμερα η κατάσταση είναι σοβαρή και αυτό το οποίο ζητούν ε, οι αγρότες ε, δεν είναι συμπόνια αλλά δικαιοσύνη. Σήμερα όμως αυτό το οποίο μας προτείνετε εσείς ε, είναι μείωση των ποσοστώσεων και είναι η αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων. Αυτά Αυτές οι δύο προτάσεις δεν δίνουν μια λύση στην κρίση. Χρειάζονται και βραχυπρόθεσμες απαντήσεις αλλά και ε, μεσοπρόθεσμες. Οι βραχυπρόθεσμες αφορούν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών όπου η κατάσταση είναι σαφής χρειάζεται μία μείωση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων έτσι ώστε να εξισορροπήσει η προσφορά με τη ζήτηση. Μείωση 5%. Δεύτερον πρέπει να ασκηθεί μία πίεση στις βιομηχανίες που συνεχίζουν να ε, δημιουργούν μεγάλους ομίλους διότι η κατάσταση δεν είναι σωστή αυτή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί να, να καθορίζουν δηλαδή τις τιμές χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το κόστος παραγωγής. Μετά χρειάζονται και μεσοπρόθεσμα μέτρα. Δεν πρέπει απλώς και μόνο να ξέρουμε ποιος παράγει αλλά και πώς παράγει και εδώ αναφερθήκατε στην Κοπενχάγη. Σήμερα όμως ο, τρόπος παραγωγής, η μο, μέθοδοι παραγωγής που χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη είναι, έρχονται σε αντίθεση με την Κοπενχάγη. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την λογική, να παράγουμε το γάλα εκτός εδάφους και να στηριζόμαστε ε, σε εισαγωγές σόγιας που έρχονται από τον Νότο αγνώντας την γεωργική παραγωγή των χωρών αυτών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την παραγωγή σε χόρτο αν θέλετε. Θα πρέπει τώρα στα, σε ένα γενικότερο πλαίσιο να ξανασυζητήσουμε ε, για τις διαπραγματεύσεις με τον, στον ΠΟΕ κάτι το οποίο δεν ε, θίξατε. Ξέρουμε σήμερα ότι το άνοιγμα των αγορών και το βλέπουμε αυτό για το γάλα και για το βόλιο κρέας για τις εισαγωγές απλώς ε, και μόνο θα αποσυντονίσουν τις δυνατότητες των γεωργών να ζήσουν και απλώς και μόνο θα, θα, θα, θα εξαφανίσουν που δεν είναι τόσο αποδοτική. Έτσι όπως ε, έκανε και το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να, ε, πριν από μερικούς ε, μήνες να επαναφέρουμε την αρχή της κυριαρχίας για τα διατροφικά θέματα όλων των χωρών του κόσμου. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να υποστηρίξω τις προθέσεις σας να καταργήσετε τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις μέχρι το 2015 και όπως είπαν και άλλοι αριστεροί αν θέλετε συνάδελφοι θα οδηγηθούμε με τον τρόπο αυτό σε μια πιο αποτελεσματική γεωργία. Εμείς αγοράζουμε 12 λίτρα γάλα κάθε εβδομάδα στην οικογένειά μου και ξέρω, παρακολουθώ από κοντά την κατάσταση ε, στο γαλακτοκομικό τομέα. Έχω μιλήσει με τους παραγωγούς και το βασικό πρόβλημα είναι πιο πόσο τους αγοράζουν το γάλα ποια είναι η τιμή του γάλακτος στον παραγωγό. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και στην τιμή πώλησης ε, στον κατελικό καταναλωτή. Ξέρω ποια είναι η κατάσταση, ξέρω πόσο δύσκολο είναι για τους παραγωγούς να πουλήσουν την παραγωγή τους ε, επιτόπου. Ε, αντιμετωπίζουν Ε, τεράστια προβλήματα στον ε, στον τρόπο διάθεση ε, του προϊόντος του. Επομένως, μήπως θα μπορούσαμε να ασκήσουμε και μία πίεση στους εμπόρους, στου μεσάζοντε. Επίσης, γιατί να μην προωθήσουμε το γάλα, γιατί είναι και θέμα ζήτησης ούτω ή άλλω. Μήπως θα μπορούσαμε να προωθήσουμε την κατανάλωση γάλατος στα σχολεία, ας πούμε θα μπορούσαμε να, ας πούμε έχουμε ούτως ή άλλως ε, στο Κοινοβούλιο δίναμε ένα καλό παράδειγμα. Σε ορισμένες ε, συνεδριάσεις προσφέραμε και γάλα. Τώρα το νερό, μονάχα νερό, καφέ και τσάι προσφέρεται. Μήπως μπορούσαμε να κάνουμε και για το γάλα κάτι. madam Dodds, please. Thank you, Mr. President. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ. Είμαι νέο μέλος από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και έχει επηρεαστεί η Βόρεια Ιρλανδία δυσανάλογα από την κρίση του γάλακτος. Πολύ απογοητευτικό γεγονός αυτό. Βεβαίως, βεβαίως, πολύ σωστό να στοχεύουμε σε μακροπρόθεσμα προγράμματα, αλλά αυτό δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα του σήμερα, τους παραγωγούς που βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση. Θα ήθελα η Κομισιόν να εξετάσει και βράχει πρόθεσμα άμεσα μέτρα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ζωοτροφές. Πρέπει να εξετάσουμε την πολιτική μηδενικής ανοχής για τα, ε, με τα τροποποιημένα προϊόντα, γενετικά τροποποιημένα προϊόντα ειδικά στις ζωοτροφές και θα θέλαμε να δούμε προτάσεις που αφορούν την αύξηση της ζήτησης για το γάλα να γίνει κάτι και προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, πολλοί μίλησαν για την ανάγκη να εξετάσουμε τα προβλήματα της διατροφικής αλυσί, της ε, αλυσίδας ε, παραγωγής, δηλαδή τι γίνεται με τις τιμές από την παραγωγή στην κατανάλωση και επίσης χρειαζόμαστε στοχευμένη χρηματοδότηση για αυτούς τους ε, παραγωγούς που βρίσκονται σε αυτή τη χείριστη θέση. Η κυρία Μόρι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω την εισαγωγή ενός μιας νέας αρχής που λέγεται Social Cross Compliance δηλαδή την κοινωνική ε, επικάλυψη συναφών μέτρων, ε, έτσι ώστε οι παραγωγοί να λαμβάνουν μία ενίσχυση όταν δημιουργούν θέσεις εργασίας. Εάν δημιουργούν θέσεις εργασίας ανάλογα με την έκταση της παραγωγικής τους μονάδας, να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση. Έχω συγκεκριμένες ιδέες και τις έχω μάλιστα και γραπτές και προθήμως θα σας τις υποβάλω. Δεύτερον, είμαι νομική σύμβουλος, είμαι νομικός εμπειρογνώμων στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι right to eat... Ε, ε, η επαρκής κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ανθρώπων είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να έχουν την εξασφάλιση ότι, ότι θα έχουν τα σωστά τρόφιμα, θα έχουν επάρκεια τροφίμων και τη σωστή ποιότητα και ότι θα μπορούν οι άνθρωποι μέσα στις κοινότητές τους να αποφασίζουν τι χρειάζονται και τι τρόφιμα επιθυμούν και τι παραγωγή θέλουν να, να αναπτυχθεί. Η παραγωγή στην Ουγγαρία με έχουν, μου έχουν τονίσει πάρα πολλές φορές ότι με πολλά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται σήμερα το φθινόπωρο ε, εκατοντάδες ε, παραγωγοί θα χρεοκοπήσουν διότι εκτός από την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν και τις χαμηλότατες τιμές ανταγωνίζονται άλλες χώρες που επιδοτούν τη γεωργία τους. Είναι λοιπόν άδικο αυτό, εκατοντάδες χιλιάδες ε, θα χρεοκοπήσουν αυτό το φθινόπωρο, διότι και οι κλιματικές, κλιματολογικές συνθήκες είναι τραγικές και έτσι οι τράπεζες που τους έχουν δανείσει θα, αναγκαστούν, θα τους αναγκάσουν να χρεοκοπήσουν και θα πάρουν πίσω τη γη που τους ανήκει. Τι θα κάνετε από αυτό. κοιτάξτε, πρέπει να βιαστούμε διότι σε πέντε λεπτά θα πρέπει να δώσω λόγο στην η κυρία Επίτροπα. Διαφορετικά θα έχουμε χρόνο. Κυρία Γέγκλα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ε, θα είμαι σύντομη. Σα ευχαριστώ που ήρθατε για την ειλικρινή σα τάση όλα αυτά τα χρόνια. Το απόγευμα θα μιλήσω επί του προπολογισμού και θα συζητήσουμε την επιστροφή εξαγωγών και ε, την παρέμβαση και πιστεύω να έχουμε θετικό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία. Αυτή τη στιγμή βεβαίως ε, είναι αναγκαστικό να το κάνουμε αυτό την, ε, τον καθορισμό των ποσοστώσεων ετησίω. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε όμως και άμεσες ενισχύσεις. Όταν λέτε ότι θα καταργηθεί η ποσόστοση το 2015. Πρέπει να έχουμε σαφεί απαντήσει στις ερωτήσεις των παραγωγών που μας ρωτάνε συνέχεια. Τι θα γίνει, τι θα γίνει και τι, τι πορεία θα ακολουθήσουμε μετά το 2015. Συγκεκριμένε απαντήσει, λοιπόν. Ήλπιζα να ακούσω ακριβώ ε, τις απαντήσεις ε, από εσά. Η άμεση ενισχύσει καλώς, αλλά μέσω πρόθεσμα τι θα γίνει μέχρι το 2015, 2015 και μακροπρόθεσμα μετά τι θα γίνει. Όσον αφορά το Ταμείο Γάλακτος, τη δημιουργία ενός έκτακτου ταμείου, αυτή η ιδέα εισήχθη ε, όταν είχαμε υπολογίσει ότι τα χρήματα αυτά μπορούν να διατεθούν. Εγώ εμπαίνω σε αυτή τη δημιουργία του Ταμείου και πιστεύω ότι είναι σωστή ιδέα. Ο κύριος Αντιπρόεδρος μας, κύριος Νικουλέσκο. και μετά ο Μπάτζη. Δυστυχώ δεν θα μπορέσει κανεί άλλο να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όπως γνωρίζουμε η σημερινή συζήτηση μονοπολήθηκε από την κρίση στον γαλακτο... γαλακτοκομικό τομέα. Αυτό δεν αποτελεί παρά ένα κομμάτι της γενικότερης κρίσης που πλήττει την γεωργία. Φυσικά σε παρόμοιες ε, περιόδους ε, χρειάζεται η παραγωγή να επιδοτηθούν και οι άμεσες ενισχύσεις που αναφέρθηκαν από την κυρία Μορβάη προ λίγο είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχει κατάσταση. Εάν οι πιο παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λαμβάνουν σημαντικές επιδοτήσεις, ε, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι νέες χώρες ε, δεν ε, λαμβάνουν τέτοιες επιδοτήσεις, τουλάχιστον όχι επαρκώς. Δεν θέλω να ξαναρχίσω την συζήτηση, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω ποιες είναι οι αλλακτικέ λύσεις προκειμένου να αποφύγουμε την περαιτέρω μείωση των παραγωγών στην Ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, η αξιοπιστία της ε, Κομισιόν, η δική σας, η προσωπική αξιοπιστία θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα των μέτρων που θα ληφθούν στον τομέα των ε, γαλακτοκομικών. Είναι σαφές, η ρύθμιση της αγοράς ε, δεν είναι ικανοποιητική, οι προτάσεις δεν ικανοποιούν και η πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα έχει αποτύχει. Κυρία Επίτροπη, είσαστε ανοιχτοί σε νέες συγκεκριμένε προτάσεις. Καταρχάς την πρόταση που υπέβαλε το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας για την αύξηση των ε, ε, ε, εξαγωγικών ενισχύσεων για κάποια γαλακτοκομικά προϊόντα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σας για την πρόταση που έκανε ο Ούγγρος Υπουργός που είχε σαν στόχο να αυξηθούν οι τιμές του ποσοστό κατά 50% διότι στο τομέα αυτό τα νέα κράτη-μέλη μετά το phasing in βρίσκονται σε χειρότερη θέση. Τρίτον, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εξισορροπήσει την ε, κυριαρχία των μεγάλων εμπορικών ομίλων και αυτό μετά από προσπάθειες, παρά τις προσπάθειες πολλών ετών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην Επίτροπο για να απαντήσει. Λυπάμαι για τους υπόλοιπους 12, 13, 15 εγγεγραμμένους στον κατάλογο των ομιλητών, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να ε, ευχαριστήσουμε και την Επίτροπο που μας έδωσε αυτό τον παραπάνω χρόνο. Ε, και μετά είναι και βεβαρημένη η ημερήσια διάταξή μας. Επίσης να υπογραμμίσω ότι και τον Ιούλιο και τώρα η Επιτροπή μας τόνισε με αποτελεσματικό τρόπο πιστεύω την ανάγκη να γίνει κάτι παραπάνω. Και σήμερα ε, ε, θα θέλαμε και θα το, θα το μεταφράσουμε αυτό και με μια πίεση που θα ασκηθεί στην Ολομέλεια του Στρασβούργου ε, δηλαδή θα υποβάλουμε μια άμεση ερώτηση προς την Επίτροπο για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπίσουμε αυτή την δραματική κρίση και όλοι πρέπει να έχουμε ένα αίσθημα ευθύνης ε, διότι μιλάμε για μια επιτροπή ε, που σε, λίγα, σε λίγες εβδομάδες ε, θα έχουμε τις ίδιες αρμοδιότητες με το Συμβούλιο. Δηλαδή, δεν θα μιλάμε μόνο, θα προτείνουμε και συγκεκριμένα μέτρα. Άρα πρέπει να είμαστε αρκετά υπεύθυνοι έτσι ώστε απλώς και μόνο να μην υπογραμμίζουμε στο μέλλον τις δυσκολίες και τα προβλήματα του τομέα, αλλά να έχουμε και συγκεκριμένες προτάσεις να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Μαριάννα, έχεις το λόγο. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω τα δυόμιση λεφτά που έχω το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, λοιπόν με το γαλακτοκομικό τομέα. Πολλοί από εμά θυμούνται την κατάσταση στο, το φθινόπωρο το 2007 όταν οι τιμές του γάλακτος έφτασαν στα ύψη και σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη ήθελαν να αυξηθεί αμέσως οι ποσοστώσεις, να αυξηθούν αμέσως οι ποσοστώσεις. Και αποφασίσαμε το 2% αύξηση. Και ανταποκριθήκαμε, αντιδράσαμε ε, πάρα πολύ γρήγορα και στην ενίσχυση της αγοράς όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο συμφωνήσαμε να γίνει αυτό το, το έλεγχος υγείας, το health check, πέρσι το Νοέμβριο και προσπαθήσαμε να, για να προσπαθήσουμε να ε, ε, διευκολύνουμε αυτήν την ομαλή προσγείωση της μελλοντική κατάργησης. αν θέλουμε τώρα να πιστοχωρήσουμε, τότε θα υπάρξει συντριβή της αγοράς το 2015. Μην ξεχνάτε ότι το σύστημα ποσοστώσεων δεν είναι υποχρεωτικό, είναι μια δυνατότητα, μια πιθανότητα, ένα, ε, μια οψιόν που υπάρχει. Και γι' αυτό έχουμε δει αυτή την αντίδραση στις χαμηλές τιμές από τον τομέα και σήμερα είμαστε 2,4% κάτω από το προϊόν. Ε, γι' αυτό ποτέ δεν θα είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να έχουμε πλειοψηφία, οι περισσότεροι δηλαδή από εμά, να ψηφίσουν υπέρ της επανεισαγωγής των ποσοστώσεων. Διότι θα δείτε μια άμεση αντίδραση από τους παραγωγούς που έχουν νόμιμες απαιτήσει και θα ζητήσουν αμέσως την επόμενη στιγμή δηλαδή αποζημίωση και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει και ούτε πρέπει να γίνει διότι είναι η εσφαλμένη κατεύθυνση. αντιδράσαμε στην κατάσταση της αγοράς από την αρχή με την εισαγωγή ιδιωτικής αποθήκευσης, ε, με την εισαγωγή της ε, ε, παρέμβασης σε πολύ πολύ ψηλότερα επίπεδα από το παρελθόν που υπήρχαν ανώτατα όρια. Επίσης, αυτή τη στιγμή διευρύνουμε, επεκτείνουμε την περίοδο παρέμβασης και χαίρομαι ιδιαίτερα που υποστηρίζει η Επιτροπή σα αυτήν την ε, επέκταση. Όσον αφορά την επιστροφή εξαγωγών βρίσκονται σε αποδεκτά επίπεδα. Δεν θέλουμε να μας κατηγορήσουν ότι διαταράσσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης των αναπτυσσομένων χωρών και γι' αυτό προχωρούμε με προσεκτικά βήματα αν και υπέστη μεγάλες πιέσεις να αυξήσω τις επιστροφές εξαγωγών τους τελευταίους 12 μήνες. Αλλά αντισταθήκαμε στις πιέσεις αυτές και δεν εξολέψαμε και τόσα κονδύλια, 174 εκατομμύρια νομίζω ευρώ στις επιστροφές εξαγωγών εκ των οποίων τα περισσότερα δαπανήθηκαν στο σύστημα παρέμβασης. Επίσης, για την κατανάλωση, για την κατανάλωση, για τη ζήτηση του γάλακτος. Ε, έχουμε κάνει πολλά βήματα και θα κάνουμε κι άλλα με ένα ειδικό ε, πρόγραμμα, μια ειδική εκστρατεία προώθησης του προϊόντος. Επίσης οι αρχηγοί κρατών και οι ε, κρατών μας ζήτησαν να λάβουμε μέτρα για τον τομέα και να απαλύνουμε την οικονομική δυσχέρεια των παραγωγών. Και για τις άμεσες πληρωμές δώσαμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να καταβάλουν τις πληρωμές στις 16 Οκτωβρίου αντί ε, στο τέλος του έτους. Επίσης προτείναμε την αύξηση του de σε 15.000 ευρώ. Επίσης προτείναμε τη δυνατότητα των κρατών μελών να, να μην εξετάσουμε το σύστημα Ποσοστό σε εθνικό επίπεδο αλλά σε περιφερειακό επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα σούπερ, μια, ένα σούπερ δηλαδή, μια, ένα ε, ε, ε, επιπλέον δηλαδή δασμός στον παραγωγό όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο για να μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο να παγώσει η ποσόστοση έτσι ώστε να επέλθει μια ισορροπία να μπορούν ορισμένοι παραγωγοί να αυξήσουν την ποσόστοσή τους ενώ σε ορισμένους άλλους που έχουν υπερπαραγωγή θα παγώσει η ποσόστοση. Ένας από τους λόγους που και πάλι πειράζει την ισορροπία προσφορά ζήτηση είναι το εξή. Αυτό που είδαμε το φθινόπωρο του 2007 είδαμε ότι ο τομέα, ο οποίο συνήθω χρησιμοποιεί προϊόντα γάλακτο στην παραγωγή, Σταμα... μείωσαν την χρήση του γάλακτος ε, και άλλαξαν προς την χρήση ε, ε, φυτικού ελαιών διότι ήταν πιο φτηνό καλαμποκιάλεο και άλλα φυτικά ελαία για την παραγωγή προϊόντων. Άρα λοιπόν δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη σε αυτό το τομέα και έχω περάσει πολλές νύχτες άϊπνοι για να βρω λύσεις που δεν θα υπονομεύσουν την κατεύθυνση που έχουμε επιλέξει. Πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε αποφασίσει μακροπρόθεσμα είναι τα σωστά για το μέλλον του τομέα. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα να σηκώσω τα χέρια ψηλά και να πω τα δέχομαι όλα, όλες αυτές τις ωραίες ιδέες ε, για να καθησυχάσω τους πάντες και να τους ευχαριστήσω. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, διότι έτσι δεν θα εκπληρώσω τα καθήκοντά μου. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι προσπαθώ να βρω, να βρω μια σωστή ισορροπία και με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω ε, λένε ότι οι, οι τιμές σταθεροποιούνται. Υπάρχει μια σταθεροποιητική τάση στις ε, τιμές ε, προϊόντων. Ε, είδαμε ότι η Φροντέρα που είναι ένας από τους μεγάλους παίκτες διεθνώς αύξησαν τις ε, τιμές τους και αυτό επηρεάζει τις τιμές διάθεσης δηλαδή στις δημοπρασίες που γίνονται και αυτό έχει μια θετική επίδραση στην αγορά. Επίσης ε, οι τιμές του βούτυρου έχουν εξελιχθεί θετικά, ιδίω στην παρέμβαση του τελευταίου μήνες είχαμε μια πολύ ψηλή προσφορά για το βούτυρο και το γάλα σε σκόνη. Βλέπω λοιπόν ορισμένα θετικά σημάδια που παρουσιάζονται στην αγορά παρέμβαση και ακριβώς αυτά είναι, ε, θα έλεγα, αισιόδοξα. Ε, θα συζητήσουμε όλα τα θέματα αυτά στο Συμβούλιο την ερχόμενη Δευτέρα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ και σε, ορισμένες, ε, σε ορισμένα άλλα ερωτήματα. On the import of, um, of soybean. Uh, I know that... Όσον αφορά τις αγωγές ε, σόγιας ε, σπόρων. GMO imports. But I think we have to keep in mind today, I would say... E- θα έλεγα ότι πάνω από 80% της εισαγωγής σόγιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γενετικά τροποποιημένη Είναι GMO. Είναι γεγονός. Αυτό είναι πραγματικότητα και δεν θα αλλάξει. Διότι βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Βραζιλία και η Αργεντινή χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τροποποιημένη σόγια. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν να τους ανταγωνιστούμε με ανταγωνιστικές τιμές στην Ευρώπη, θα σκοτώσουμε θα εξοντώσουμε τη δική μας παραγωγή κρέατος. Διότι τι θα συμβεί αν θέλουμε να κάνουμε εισαγωγή ε, αποκλειστικά μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων ή προϊόντων με, μηδενική, με μηδενικό ποσοστό ανοχής δεν λέω ας πούμε το 0,5 ποσοστό ανοχής ή κατόφλι για μη εγκεκριμένα GMO προϊόντα. Εμείς τεχνικά χρειαζόμαστε 0 ποσοστό. Διαφορετικά θα, θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στο τομέα κρέατος. Εάν λοιπόν εξετάσετε το σενάριο που θα πρέπει πρέπει να εισάγουμε ε, μη τροποποιημένα προϊόντα ή μόνο προϊόντα με ένα πάρα πολύ χαμηλό κατόφλι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον τομέα του κρέατος και τι θα γίνει. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε εισαγωγή ε, ε, βοηδών η εισαγωγή κρέατος από άλλα μέρη του κόσμου και ξέροντας όμως ότι τα ζώα αυτά ή τα προϊόντα αυτά έχουν τραφεί με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές. Οπότε τελικά τι θα κάνουμε, θα εξαπατούμε τους καταναλωτές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ε, διαφανή πολιτική εγώ δεν υπεραμείνουμε τις αποδυνάμωσης ε, της πολιτικής μας, αλλά προσπαθώ να βρω και μέτρα που δεν θα εξοντώσουν τον τομέα της, ε, του κρέατος. Όσον αφορά τις μπανάνες και τις ντομάτες, όταν συμφωνήσαμε για τις μπανάνες και συμπεριλάβαμε την ενίσχυση της ε, μπανάνας, ήταν μια χρυσή λύση αυτή για τους μπανανοπαραγωγούς. Χρυσή λύση τους χρυσώσαμε. Έχουμε τώρα, διαπραγματευόμαστε με τις χώρες ΑΚΕ και δεν ξέρω αν θα βρούμε λύση, αλλά θα κάνουμε μία αναθεώρηση της πολιτικής μπανάνας και αυτό είναι μέσα στην ατζέντα μας. Και αναφέρεται και στα συμπεράσματα μάλιστα ε, αυτού του θέματος. Για τον ΠΟΕ, αύριο το πρωί θα πάμε στο Νέο Δελχή για να συναντήσουμε 35 υπουργού εμπορίου κυρίω από τις αναπτυσσόμενες χώρες διότι θέλουν να προωθήσουν τις συζητήσεις αλλά και την, ε, τα συμπεράσματα για τις ε, διαπραγματεύσεις στο ΩΣΑ και ε, μετά από τις συναντήσεις των G8 να ολοκληρωθούν τα ντοσιέ το, οι προτάσεις μας υποβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2008. Τότε είχαμε ένα πολύ στενό διάλογο με το Συμβούλιο και το Συμβούλιο ήταν, ήταν παρόν τότε σε όλες τις διαπραγματεύσεις και προφανώς βεβαίως αυτό το, αυτές τις προτάσεις θέλουμε να ολοκληρώσουμε του 2008. Ο Ζωζέ Μποβέ ανέφερε την μείωση των ποσοστών γάλακτος. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα, απλώς θα πω ότι για την παραγωγή πρωτεϊνών στην Ευρώπη είναι, είναι δυνατόν για τα κράτη-μέλη μέσω του άρθρου 68 να βελτιώσουν τις ενισχύσεις τους για αυτές τις καλλιέργειες. Και ξέρω ότι η Πολωνία και η Γαλλία θα χρησιμοποιήσει αυτές αυτή τη δυνατότητα το άρθρο 68. Το θέμα της ανισορροπίας μεταξύ ε, της ανισορροπίας των, των ε, αμέσων πληρωμών μεταξύ νέων και παλαιών κρατών αυτό το θέμα θα συζητιέται στο μέλλον για το μέλλον της ε, ΚΑΠ μετά το 2013. Όταν, κάναμε αυτό τον, όταν συμφωνήσαμε για τον έλεγχο υγείας είχε γίνει μία δήλωση από όλα τα κράτη-μέλη ότι δεσμεύονται, ότι θα δεσμευτούμε για να βρούμε μία σωστή λύση για την κατάργηση αυτής της εξομάλυνση μάλλον αυτής της ανισορροπίας. Πρόεδρε, αυτά είχα να πω και δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ περισσότερο το χρόνο σας. Όπως ξέρετε είμαι πάντα πρόθυμη να επιστρέψω και να συζητήσουμε μαζί τα θέματα που σας, σας ενδιαφέρουν. Ε, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας και θα τα ξαναπούμε στις 15.00 για να συνεχίσουμε τις αρχές της Επιτροπής. Γεια σας. Yes.